Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και καλώς ήρθατε σε αυτήν την ε, έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλωσορίζουμε επίσης και τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκι. Ευχαριστούμε πολύ και εσείς που ήρθατε τόσο νωρί σήμερα το πρωί για τον διαρθρωμένο μας διάλογο. Υπό την ιδιότητά σας, Αντιπροέδρου υπεύθυνου για την οικονομική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ένωση κεφαλαγορών. Να κρίνουμε την ημερήσια διάταξη πρώτα απ' όλα. Συμφωνείτε? Ωραία. Και συνεχίζουμε και περνάμε στο διαθρωμένο μας διάλογο, ο οποίο έχει να κάνει, όπω είπαμε, με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και ένωση αγορών. Όπω γνωρίζετε, ο αντιπρόεδρο Νταμπρόφσκης επίση θα πάει στις 10 Δεκεμβρίου μαζί με τον Επίτροπο Μοσκοβίση ε, στην, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Έτσι και αλλιώς ήταν απόφαση και των συντονιστών υπό το άρθρο 7.3 του κανονισμού του ΠΑΚ. για τη γνωμοδότηση όσον αφορά τον Ιταλικό προπολογισμό. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε λοιπόν σήμερα. Και στόχος μας είναι να επικεντρωθούμε στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Κάνουμε πολύ καλή δουλειά, εντατικά εργαζόμαστε για να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται ε, μεγαλύτερο κομμάτι των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημειώνουμε επίσης ότι χτες είχαμε δύο ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που σημειώνουν τις ε, τελευταίες, ε, τα τελευταία νέα σε σχέση με την μείωση του κινδύνου και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης θέλω να σας πω ότι χτες συνεδρίασαν οι σκιώδεις εισηγητές, οπότε στις 6 θα ψηφίσουμε, αυτό επιβεβαιώθηκε. Συνεπώς προχωρούμε πολύ γρήγορα και για αυτές τις προτάσεις. Και όπως λέει και η ανακοίνωσή σας, ενθαρρύνουν τα στοιχεία, επιταχύνονται οι διαδικασίες και θα μπορέσουμε έτσι να τα καταφέρουμε με το ρυθμιστικό πλαίσιο και το backstop. Βέβαια, στόχος μας είναι να εγκρίνουμε και τα δύο νομοθετικά κείμενα. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε διαδικασία fast track για τον κανονισμό δεν σημαίνει ότι δεν θα προχωρήσουμε και με την οδηγία. Ζητούμε και από το Συμβούλιο να κάνει το ίδιο για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε, ακόμα και αν δεν προχωρούμε παράλληλα, ε, να προχωρήσουμε και με τα δύο στοιχεία του πακέτου για τον κανονισμό και την οδηγία. Ακόμα δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση, αλλά τύπα υπάρχει συμφωνία για το τραπεζικό πακέτο και ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Έγινε πάρα πολύ δουλειά. Εμείς επιταχύναμε άνευ προηγουμένου τις διαδικασίες για να βοηθήσουμε με τη δικιά μας πολιτική συνεισφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και ελπίζουμε ότι και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επιδείξει την ίδια φιλοδοξία. Αλλά πολύ μίλησα. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης για τις δικές του εισαγωγικέ παρατηρήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Άξιο τιμή, ευρωβουλευτέ, ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να έρθω σήμερα και να απευθυνθώ σε εσά. Όντω, το οικονομικό κλίμα δεν ε, καλύπτεται από βεβαιότητα, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι δυνατή, να μπορεί να αντιμετωπίσει τις διάφορες, τους διάφορους τριγμούς. Σημαίνει ότι πρέπει να διατηρήσουμε τις ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές μας αγορές, να είναι ανθεκτικές σε σοκ Πρόσφατα επιταχύθηκαν οι διαδικασίες για νομοθεσία, όπως μας είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής. Έρχονται όμως και οι ευρωεκλογέ τις επόμενες εβδομάδες λοιπόν, και μιλάμε για εβδομάδες πιο όχι για μήνες, πρέπει να προχωρήσουμε για να πετύχουμε την αναγκαία πρόοδο. Χτες λοιπόν εγκρίναμε δύο εκθέσεις πρόοδου για την Τραπεζική Ένωση και τις αγορές και θέλω να σας μιλήσω ακριβώς για την πρόοδο αυτή και επιπλέον θα πω και δύο λόγια για το FinTech. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, οι χθεσινές εκθέσεις δείχνουν ότι προχωράμε, ότι η χρηματοστική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενισχυθεί. Όμως, ακόμα υπάρχουν θύλακες αδυναμίε. και γι' αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στο νομοθετικό πακέτο τη άνοιξη για να μειωθούν τα μη ξυπηρετούμενα ε, δάνεια. Επίσης, ε, για το backstop σήμερα θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πιέσει του συνομοθέτε να έχουν καταλήξει μέχρι τα τέλη τη χρονιάς. Πρέπει όμω να θυμόμαστε για τι δευτερογενείς αγορές. Προχωρούμε επίση, και αυτό αποτελεί κομμάτι του πακέτου. Το Prudential Backstop λοιπόν γίνεται, προχωράει. Επίσης, αυτό που είναι καλό είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία σε σχέση με το πακέτο το τραπεζικό για το, του 2016. Και στον τριμερή διάλογο προχωρούμε. Το πακέτο αυτό σίγουρα θα προσφέρει μεταρρύθμες και θα προσαρμοστεί σε διεθνή πρότυπα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένη της πρόοδου που έχει γίνει, ζητάει να υπάρξει και για τον ΙΜΙΕΣ μια συμφωνία ενιαία και να ακολουθήσουμε και άλλα βήματα για τις εγγύσεις καταθέσεων. Και εδώ ζητούμε στις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις και να διασφαλίσουν το έντις ότι θα προχωρήσει. Έρχομαι τώρα στην ε, Ένωση Κεφαλαιογορών. Και εδώ ε, πρέπει να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν οι αποταμιεύσεις για περισσότερες επενδύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τις διάφορες νομοθετικές προτάσεις θέλουμε την Ένωση Κεφαλαιαγορών και λείπουν ακόμα 10 στοιχεία που βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ξέρω ότι εσείς δουλεύετε σκληρά για να προχωρήσετε διάφορους φακέλους, αλλά τις επόμενες εβδομάδες σας παρακαλώ να προχωρήσετε σε συμβασμούς για να επιτευχθεί πρόοδος θα υποφεληθούν πολύ και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και επενδυτές. Για παράδειγμα, για συνταξιδιωτικά προϊόντα, για να έχουν περισσότερες επιλογές οι πολίτες και με χαμηλότερο κόστος. Έχει γίνει πρόοδος, αλλά χρειάζεται παραπάνω δουλειά. Για να διασφαλίσουμε ακριβώς την πανευρωπαϊκή σχέση του προγράμματος. Επίσης, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που ζητούν οι περισσότεροι επενδυτές να επενδύσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχει η πρότασή μας για το SME, για τις μικρομεσαίες δηλαδή επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορούν να υπάρξουν ε, securities στην αγορά αυτή. Ξέρω ότι είσαστε επικοδομητικοί και ελπίζουμε αρχές Δεκεμβρίου να έχουμε αποτελέσματα. Επίσης, για τα καλυμμένα ομόλογα. Και εδώ πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε περισσότερα στην πραγματική αγορά. Το Συμβούλιο έχει συμφωνήσει, οπότε ο τριμερής διάλογος φαντάζομαι ότι μπορεί να ξεκινήσει. Όπως υπόθηκε ήδη, το Brexit ε, μας αναγκάζει να προχωρήσουμε με ακόμα πιο ταχύς ρυθμούς για την Ένωση Κεφαλαγορών. Θα αρχίσουν τριμερείς διάλογοι για τους νέους κανόνες, έτσι ώστε να υπάρχει εποπτεία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν τη νέα εποχή. Και ελπίζω να επιτευχθεί και πρόοδος όσον αφορά και την εποπτεία των επενδύσεων. Και ζητούμε τη δικιά σας στήριξη. Θέλουμε και έγκριση της αναθεωρημένης μεταρρύθμισης για τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, όπως λέει και η εντολή μας. Εδώ πέρα πρόκειται για δύο στοιχεία. Ενισχύεται η εξουσία του Ίσης που είναι κάτι πολύ σημαντικό δεδομένου του Brexit, αλλά επιπλέον ενισχύει και το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δικιά σας στάση και σας ενθαρρύνω να επιταχύνετε για να ολοκληρωθεί το έργο σας έγκαιρα και να μπορέσουν και εδώ οι τριμερείς διάλογοι να ξεκινήσουν το Δεκέμβριο. Όσον αφορά τώρα τη, τα βιώσιμα δημοσιονομικά, μετά τη Συμφωνία των Παρισίων, Έχουμε τρεις νομοθετικές προτάσεις για τα βιώσιμα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να υπάρξει περισσότερη ροή χρήματος στην αναμονημένη οικονομία μας. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να επενδύσουμε περισσότερο σε ό,τι είναι πράσινο και να υπάρξουν οι κατάλληλες προδιαγραφές και πρότυπα για μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για την πρόοδο που έχει επιτύχει μέχρι τώρα και ελπίζουμε οι συνομοθέτες μέσα σε αυτή τη θητεία να καταφέρουν να εγκρίνουν τους σχετικούς φακέλους. Παίρνω τώρα στο φίντα και τις πληρωμές. Εμείς περιμένουμε διάφορα στοιχεία ακόμα από το ΙΣΙΣ και σε συντονισμό με το έργο που γίνεται σε διεθνές επίπεδο, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο χρειάζεται ρυθμιστική δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Στο μεταξύ προσπαθούμε να πετύχουμε πιο φτηνές και καλύτερε υπηρεσίε πληρωμών για τους Ευρωπαίου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνουμε κυρίω για την άνοιξη τη ρύθμιση για τι διασυνοριακέ πληρωμές να γίνονται ε, σε ευρώ εξίσου φτηνά όπως γίνονται και μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε κάτι στις 5 Νοεμβρίου και ελπίζουμε ότι οι εταίροι θα πετύχουν κάποιο συμβιβασμό. Το ευρώ θα είναι το νόμισμα σε λίγο όλων των χωρών μελών και θέλουμε να ενισχύσουμε το διεθνή του ρόλο. Συνεπώς είμαστε πεπισμένοι ότι η θέση μας να επικεντρωθούμε στις πληρωμές μόνο σε ευρώ είναι και ο σωστός δρόμος για να προχωρήσουμε. Τέλος, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες θα οδηγήσουν σε περισσότερη ολοκλήρωση αλλά και σε καλύτερα ρυθμισμένες χρηματοπιστωτικές αγορές και θα υιοθετηθούν οι ρυθμίσεις αυτές από όλες τις επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας σε όλους αυτούς τους φακέλους μέχρι τώρα, όπως επίσης και για τη στήριξή σας τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ γενικότερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνεχιζόμενη στήριξη. Σύμφωνα βέβαια και με την θεσμική σας εντολή στον τριμερή διάλογο για τη διευκόλυνση συμφωνιών μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Βεβαίως σημειώνουμε επίσης την έκκλησή σας να δείξουμε εμείς τη μέγιστη δυνατή συμβιβαστική διάθεση. Τώρα αυτό χρειάζεται ιδίω να το δείξει το Συμβούλιο, διότι σε ορισμένα σημεία προσεγγίζουμε πλέον στη συμφωνία, όπως είναι και εδώ εισηγητής για τα BEPS και μιλήσαμε χθε και για το REFIT και βλέπουμε ωστόσο ένα δισταγμό από την πλευρά του Συμβουλίου να προχωρήσει και Ως γνωρίζετε, για να χορέψει κανείς ταγκό χρειάζονται δύο. Άρα πρέπει και το Συμβούλιο να κατανοήσει ότι ε, υπάρχουν δύο συνομοθέτες και να μετακινηθεί και αυτό από τις θέσεις του, όπως το κάνουμε και εμείς, όντας ρεαλιστές. Ας αρχίσουμε με τους αγοριτές. Και πρώτος ο Μάρκος Φέρμπερ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Καλημέρα και σε εσά κύριε Αντιπρόεδρε δύο ζητήματα με απασχολούν. Πρώτον, το Brexit Contingency Plan, δηλαδή τι γίνεται ως εναλλακτική, τι υπάρχει ως εναλλακτική λύση για την Βρετανική αποχώρηση. Παρακολουθούμε μεγάλη προσοχή την εξέλιξη στην Βουλή των Κοινοτήτων και τη συζήτηση που διεξάγεται εκεί, διότι οι πιθανότητε να υπάρξει το λεγόμενο σκληρό Brexit φαίνεται να αυξάνονται πάλι. Το ερώτημα είναι τι κάνετε εσείς για να αντιμετωπίσετε ένα ενδεχόμενο τέτοιο σενάριο για τα ντοσχεία εκείνα που είναι σημαντικά για το Brexit. Όπως α πούμε η επανεξέταση, το review δηλαδή των ε, επενδυτικών εταιριών. Όλα αυτά είναι αναγκαίο να γίνουν πριν τελικώς να υπάρξει το Brexit. Το δεύτερο, Solvency 2. Πρόσφατα αρχίσατε διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση για την σχετική κατεξουσιοδότηση πράξη. Εμείς έχουμε βάλει προτάσεις. Ένα ζήτημα που μου φαίνεται σημαντικό είναι κίνητρα για μακροπρόθεσμες παραγωγικές επενδύσεις. Αυτό έχει περιληφθεί μεν στον προβληματισμό σας, αλλά βάζετε μία δωδεκαετή περίοδο και ένα ring fencing. Με τέτοιο τρόπο που στην ουσία η προσπάθεια αυτή δεν θα έχει καμία ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Πρόκειται να τα επανείδεται αυτά πριν τελικώς να εγκριθεί η κατεξουσιοδότηση πράξη. Ευχαριστώ. Ορίστε κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτα, για τον σχεδιασμό, για τα διάφορα ενδεχόμενα του Brexit. Πράγματι, πρόκειται για κάτι το οποίο λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη στις 13 Νοεμβρίου δημοσιεύσαμε το σχετικό σχέδιο Brexit Contingency Plan που περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για την ετοιμότητα και για το έργο του σχεδιασμού αυτού για το ενδεχόμενο να μην υπάρξει συμφωνία Brexit. Εκ παραλλήλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί τους διάφορους κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε σχέση βέβαια με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου κάνουμε την ανάλυση με εισρωές και από άλλα θεσμικά όργανα και έχουμε και τεχνική ομάδα εργασίας Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και Τράπεζας της Αγγλίας, οι οποίοι επίσης επεξεργάζονται τα θέματα αυτά. Και ένα από τα θέματα που ανέκυψαν ως ενδεχόμενος κίνδυνος αφορά τους συμψηφισμούς το ενδεχόμενο μείωση δηλαδή των συμψηφισμών, reduced clearing. Και γι' αυτό τονίσαμε εμεί ότι στην περίπτωση αυτή θα καταθέσουμε μέτρα για προσωρινό καθορισμό για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό. Υπάρχουν και άλλοι τομείς που συζητούνται, για παράδειγμα για τα ε, παράγωγα, και για ορισμένα θέματα ασφαλιστικής, ε, ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Αυτά τα ζητήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ωστόσο και από αυτούς που συμμετέχουν στις αγορές. Εν πάση περιπτώσει παρακολουθούμε την κατάσταση, εργαζόμαστε μαζί με τα άλλα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα και είμαστε έτοιμοι να δράσουμε εάν τελικώς υλοποιηθεί το σενάριο της ε, αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Όσον αφορά την Solvency 2. Επ' αυτής διεξάγονται εντατικές συζητήσεις και ένα στοιχείο βέβαια είναι και το ερώτημα πόσο, πόσα μπορεί κανείς να αλλάξει μέσα σε μια κατεξουσιοδότηση πράξη όταν πρόκειται για νομοθεσία επίπεδου 1. Διότι βέβαια η κατεξουσιοδότηση πράξη δεν μπορεί να αποκλίνει από το ουσιώδες περιεχόμενο της νομοθεσίας. Αυτό είναι σαφές. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να είναι σαφές ότι τα περιθώρια λιγμών εν προκειμένου είναι περιορισμένα. Ταυτόχρονα έχουμε σημειώσει και κάποιες ανησυχίες της Επιτροπής σας, Επιτροπής Οικονομικών, και όχι μόνο πρόσφατα αλλά και από παλαιότερα έτη. Για παράδειγμα, το θέμα της μεθοδολογίας που αφορά την ΕΟΠΑ για τα risk-free rates και μετά από έτοιμα δικό σας περιλαμβάνουμε και την μεταχείριση της long-term equity. Έχουμε βάλει και, και ε, εφαρμογή. Και ζητούμε από τις επιχειρήσεις να είναι προετοιμασμένες και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε μετοχές. θα χρησιμοποιήσουμε τους στόχους του CMU και ένας από αυτούς τους στόχους είναι να δοθούν κίνητρα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εξυπηρετούν ή και που είναι επενδυτές και ταυτόχρονα οφείλουν να διατηρήσουν επαρκές επίπεδο προστασίας των μετόχων. Εσείς μας ζητήσατε σημαντική μείωση του παράγοντα σοκ για τις μετοχές στη τάξη του 22%. Αυτό μπορεί ωστόσο να δικαιολογηθεί μόνο εάν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο ασφαλιστής μπορεί να διατηρήσει τις equity investments και σε περίπτωση ελέγχου stress. Και αυτό μεταφέρουμε εμείς πλέον σε νομοθεσία, αυτή δηλαδή την οικονομική λογική. Η νέα κατηγορία long term equities αποτελεί στην πραγματικότητα επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ενότητας αυτής για τις ε, μετοχές και θα ισχύει όχι μόνο για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά θα χρειαστούν και κάποιες περιορισμένες προσαρμογές, ώστε οι διατάξεις αυτές να μπορούν να εφαρμόζονται και σε άλλου είδους επιχειρήσεις και όχι μόνο στα συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάνοντας αυτό βέβαια πρέπει να διατηρήσουμε και το επίπεδο δέωσας επιμέλειας. Και αυτό θα επανέλθει το 2020 στην επανεξέταση της Solvency 2. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Υπενθυμίζουμε ότι η συνθήκη δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με την κατεξουσιοδότηση με πράξης, χωρίς όμως να γίνονται ουσιώδεις μεταβολές. Άρα βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια της βάσης της συνθήκης και εξετάζουμε προσεκτικά την απάντησή σας, αλλά εκ πρώτης όψεως η ανάγνωση που κάνουμε δεν είναι θετική, διότι η συνθήκη δίνει ε, την εξουσία στο Κοινοβούλιο να απορρίψει την ε, στην πράξη. Θα συνεχίσουμε τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίω. Η Περβάνς Μπερές έχει το λόγο. Κύριε Αντιπρόεδρε, μιλήσατε για το Brexit. Θα ήθελα να επανέλθω σε δύο πτυχές. Καταρχάς, όσον αφορά τα, τα ταμεία Ξέρετε ότι είμαι διστακτική όσον αφορά τη δυνατότητα της ισχύουσας νομοθεσίας να διατηρήσει το επίπεδο απαιτήσεων που ορίσαμε στο πλαίσιο της ΜΥΦΙΤ και της ΜΥΦΙΡ. Μη, δεν θεωρείτε ότι είναι επίγουν να ορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να εκτελεστεί αυτή η νομοθεσία για τα επενδυτικά εβάσματα γνωρίζοντας ότι κινδυνεύουμε να κενώσουμε περιεχομένου τη λογική της νομοθεσίας μη feed μη από τη μια πλευρά και από την άλλη κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουμε τη βάση για ένα καταστροφικό dumping μέσα στην εσωτερική αγορά. Δεύτερη παρατήρηση σε σχέση με το Brexit. Θα θυμάστε ότι είχαμε ε, ε, ανανεώσει τις αντιστοιχίες με το ελβετικό χρηματιστήριο για ένα χρόνο μέσα σε ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο. Αυτή η αντιστοιχία ολοκληρώνεται ε, μέσα στο τρέχον έτος. Ποια είναι η προοπτική για ανανέωση και ποια είναι και τα στοιχεία της πολιτικής συζήτησης γύρω από την ενδεχόμενη αυτή ανανέωση. Άλλη παρατήρηση. Σε μια συζήτηση στην Ολομέλεια παρατηρήσατε μια πολύ έντονη κινητοποίηση του σώματος γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Είναι σίγουρα πολύ αργά για να κάνουμε οτιδήποτε, αλλά όλο ένα και περισσότερες φωνές ε, ακούγονται και λένε ε, ότι πρόκειται για ένα πραγματικό Far West. Τι θα κάνετε ώστε η Ευρώπη να μην ε, πιαστεί πάλι απροετοίμαστη. Και έπειτα δεν αναλάβατε ευθύνες νωρίτερα για να εξεταστούν με σωστό τρόπο οι συνθήκες ε, προετοιμασίας των πρίψης στα ΕΜΠΕΜ και επιτρέπεται σε αυτά να συνεχίσουν την πίεση όσον αφορά την εξαίρεση για την εφαρμογή των πρίψη με το κίνητρο με την δικαιολογία μάλλον ότι η έναρξη ισχύω αυτή τη νομοθεσία καθυστέρησε από τον νομοθέτη όταν επρόκειτο να υιοθετηθούν οι πράξης πράξει ε, επίπεδο 2 και αυτή τη στιγμή ορισμένοι ανησυχούν για τι συνθήκε προστασία των καταναλωτών. Uh, okay. Ε, thank you much. Σας ευχαριστώ. αρκετά τα ερωτήματά σας, να μιλήσω για την αναθεώρηση, για την αναθεώρηση των επενδυτικών ταμείων. Εδώ είχαμε την υποστήριξη της Επιτροπής ΕΚΟΝ και συμμεριζόμαστε μαζί σας την μέρημνα για να εξασφαλίσουμε την προστασία για τους κεφαλαϊκούς κινδύνους αλλά και για να εξασφαλίσουμε τη γενική συμμόρφωση και να προωθήσουμε τον ανταγωνισμό είναι οι συστημικά σημαντικές επενδυτικές εταιρείες που ασκούν και τραπεζικές δραστηριότητες θα πρέπει να θεωρούνται ως πιστοτικά ιδρύματα και να ρυθμίζονται και να εποπτεύονται πλήρως όπως και οι τράπεζες. Η πρόταση της ΕΚΟΝ για να μπορέσουν οι αρμόδιες αρχές να ορίσουν άλλες εταιρείες που εκθέτουν που παρουσιάζουν μάλλον τραπεζικούς ε, ε, κινδύνους να παραμένουν στο CRD ε, συζητιέται σε, μέσα σε τριμερούς, τριμερείς διαλόγους με κράτη-μέλη που θέλουν να διατηρηθούν όλοι αυτοί στο CRD. Όσον αφορά και τις αλλαγές στις αγορές στο MIFID και MIFIR, Θεωρούμε πως ίσως οι προτάσεις της ΕΚΟΝ είναι υπερβολικές. Ίσως να χρειαστεί στοχευμένη νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε ανοιχτοί για να το συζητήσουμε με επικοδομητικό τρόπο. Επίσης πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η Ευρώπη να μην εξαρτάται από ε, εταιρείε τρίτων χωρών για επενδυτικέ ε, υπηρεσίες. Για την Ελβετία τώρα έχουμε ε, εγκρίνει προσωρινή αντιστοιχεία για ένα χρόνο για τα χρηματιστήρια σύμφωνα με το ΜΥΦΙΡ. Και φέτος ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία. Στην προσέγγιση μας βασικά ακολουθούμε το παρίσματα του Συμβουλίου που ε, επαναλήφθησαν δις και ορίζουν ότι η προϋπόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη της τομεακής προσέγγισης παραμένει η θέσπιση ενός κοινού θεσμικού πλαισίου. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πόσο γρήγορα η Ελβετία μπορεί να κινηθεί προς ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο. Αυτό είναι το θέμα κλειδί πράγματι παρέμβαση της κυρίας Μπερές εκτός μικροφώνου. Ε, ο κύριος Δομπρόφης συνεχίζει. Εξαρτάται εάν θα υπάρξει πρόοδος με το πλαίσιο ισοτιμίας. Ε, αν δεν υπάρξει, θα εκπνεύσει η ισχύουσα ε, ισοτιμία. έτσι έχει η κατάσταση. ναι, αλλά έχουμε μόνο μία ώρα, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, λακωνικά. Για τα ΠΡΙΠ αναμένουμε ότι θα ολοκληρώσει το ρυθμιστικό χάρτη τον επόμενο μήνα. Α, για τα κρυπτονομίσματα, με συγχωρείτε. Ε, θα αν όντω ολοκληρωθεί αυτό τον επόμενο μήνα, θα αποφασίσουμε τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την ε, χρήση και τον ΠΡΙΠ, στόχος μας παραμένει να εξασφαλίσουμε την συμβατότητα για όλα τα προϊόντα λιανική. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε στην παράταση και στην επέκταση των USIT, αλλά θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο σύντομα. σε ευχαριστώ. Πρέπει να είμαι στο Ολομέλεια στις 9 γιατί θα μιλήσουμε για το Brexit. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ λακωνικοί όλοι. Η Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Καλημέρα κύριε Επιτροπέ. Ο ίδιος ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην απροθυμία του Συμβουλίου να προχωρήσει σε συμβιβασμούς σε διάφορους τομείς. Και εγώ θα πάω ακόμα πιο μακριά. Παρατηρώ ότι όλο και περισσότερο το Συμβούλιο Συνομοθέτης δεν λειτουργεί. Παρατηρείται μια δυσλειτουργία. Το είπατε και εσείς με το FinTech. Είμαστε στη μέση τριμερών διαλόγων ε, για το ΠΕΠ και έχω την αίσθηση ότι όχι μόνο εδώ, αλλά για πολλά άλλα ζητήματα αυτό δημιουργεί πρόβλημα και αποτελεί και μια απειλή στην εσωτερική αγορά. Οι στόχοι που θέλετε εσείς να πετύχετε κινδυνεύουν. Και αναρωτιέμαι γιατί προχωράμε, εκπονούμε νέα νομοθεσία, νέους κανόνες. Είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, αλλά ακόμα και όταν έχει εγκριθεί η νομοθεσία, στη συνέχεια πρέπει να τίθεται και σε εφαρμογή στις χώρες μέλη. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα ε, στους εθνικούς επόπτες, ε, για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουν και εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό επίσης υπονομεύει την εσωτερική αγορά και αποτελεί και απειλή για την δικιά μας θέση ανά τον κόσμο. Πρόσφατα διάβασα εκθέσεις για την θέση των πλατφορμών ε, ίντερνετ και φαίνεται ότι το μερίδιο των ευρωπαϊκών, και αυτό έχει να κάνει και με το FinTech, έχουν μόνο 12% του συνόλου και μόνο 2% όταν πρόκειται για την αξία στην παγκόσμια αγορά. Οπότε αυτή η απροθυμία του Συμβουλίου και των χωρών ε, μελών, η απροθυμία που είναι αυξανόμενη για την ε, ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, απειλεί τη θέση μας στον κόσμο. Οπότε αναρωτιέμαι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φροντίζει να το εξηγήσει καλά αυτό το πρόβλημα και να αντιμετωπίσει αυτό το συμβούλιο ώστε και ρυθμιστικά και χρηματοπιστωτικά. Δεν θα προλάβουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι, έχετε ξεπεράσει το λεφτό σας, οπότε κάντε την ερώτησή σας γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Τι κάνει η Επιτροπή γι' αυτό, αν είναι αρκετά προδραστική απέναντι στο Συμβούλιο. Απάντηση. Ας δούμε λίγο την πτυχή της ε, εφαρμογής ε, του ανοσιακού δικαίου και νομοθεσίας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ακριβώς έχουμε την αναθεώρηση για την Ευρωπαϊκή Εποπτεία, έτσι ακριβώς ώστε να εφαρμόζεται περισσότερο ομοιόμορφα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από τους εθνικούς επόπτες. Υπήρξαν και πρόσφατες τροποποίησεις όσον αφορά τις απαιτήσει ε, και την καταπολέμηση της νομοποίησης ε, ε, παράνομου χρήματος, με το MRL και με άλλα. Αλλά όπως είπαμε, σε εθνικό επίπεδο γίνεται η εφαρμογή. Ελάχιστες είναι οι αρμοδιότητες σε αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά το τι κάνουμε με το Συμβούλιο, συνεργαζόμαστε στενά και με το Συμβούλιο και ζητούμε από το Συμβούλιο να προχωρήσει, να προχωρήσει σε συμβιβασμούς και να υπάρξει πρόοδος για όλους αυτούς τους φακέλους που συζητάμε μέσα στην εντολή αυτή, σε αυτή τη θητεία. Γιατί οι συνομοθέτες είναι αυτοί που αποφασίζουν στο τέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως ρόλο να διευκολύνει, να δίνει πληροφορίες, αλλά τις αποφάσεις τις παίρνουν οι συνομοθέτες, δεν τις παίρνει κανένας άλλος. Ευχαριστώ εσείς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αρχίσω ε, επενώντας σας για τα πολύ σημαντικά που κάνετε για την βιώσιμη χρηματοδότηση. Εργαζόμαστε και εμείς σκληρά από πλευράς του Κοινοβουλίου με τρεις νομοθετικές προτάσεις που μας έχετε διαβιβάσει. Αντιλαμβάνομαι ότι για την ταξονομία αυτό που θέλετε είναι να δείτε ποιο είναι, τι πράγμα είναι βιώσιμο και είναι σημαντικό να δει κανείς και τι λένε οι ειδικοί και για το περιβάλλον αλλά και για τα οικονομικά χρηματοδοτικά. Δεν έχουμε προτάσεις όμως για αποκλεισμένους τομείς. Ίσως θα μπορούσε ένα πράσινο ομόλογο να περιλάβει για παράδειγμα και θέματα ε, καυσίμων κλπ. Η ερώτησή μου είναι, συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η τελική νομοθεσία δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζει ποια οικονομική δραστηριότητα είναι βιώσιμη αλλά και πια δεν είναι βιώσιμη και να οδηγηθούμε τέλος σε παραμερισμένα στοιχεία ενεργητικού. Σε μια όμως μετάβαση, αλλά να δώσουμε ξεκάθαρα σημεία, ξεκάθαρα σημάδια δηλαδή μηνύματα στην ε, βιομηχανία, αλλά και ξεκάθαρες προθεσμίες. Ναι, Ευχαριστώ. Πρόκειται για ερώτηση για τη λεγόμενη καφετιά ταξονομία, brown taxonomy. Και κάτι το οποίο εξετάζουμε πριν να καταθέσουμε την νομοθετική μας ε, πρόταση για την ταξονομία. Ε, είπαμε πράσινη ταξονομία, καφετιά ταξονομία. ώστε να είναι λιγότερη περίπλοκη νομοθεσία αυτή. Γι' αυτό προτιμήσαμε να ξεκινήσουμε από την πράσινη ταξονομία, την οποία θα χρειαστεί να αναπτύξουμε σταδιακά, βαθμιδών. Ξεκινούμε λοιπόν, όπως ξέρετε, με μέτρα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, που περιλαμβάνονται και άλλες πτυχές, και βλέπουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία που εξελίσσεται, σχετικά δηλαδή με το τι θεωρούμε πράσινο και τι όχι, και θα αναπτυχθούν σχετικώς οι, οι ταξονομίες. Για την ώρα νομίζουμε ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Όπως είπα, για να υπάρχει μια πιο απλουστευμένη προσέγγιση. Μπορούμε ίσως να βάλουμε και κάποια στοιχεία για τις μελλοντικέ καστανές, ας το πω έτσι, ταξονομίες, αλλά δεν το κάνουμε ακόμη, διότι ειλικρινά δεν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο θα περάσει από το Συμβούλιο. Οι τρέχουσε προτάσει ήδη αντιμετωπίζονται με κάποια επιφύλαξη από κάποιο δισταγμό από το Συμβούλιο και θέλουμε σε πάση περιπτώσει να προχωρήσουν. Μπορείτε να μου δώσετε ένα λεπτό ακόμα για να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε για το Συμβούλιο και είναι σημαντικό όντω να συμφωνήσουν και αυτοί η ανησυχία μου όμω, όπω είπα και στην ερώτηση, είναι ότι ίσω καταλήξουμε σε μια κατάσταση όπου θα έχουμε ένα ορόσημο, ένα benchmark και πράσινο ομόλογο και μέσα σε αυτό θα μπουν και βιομηχανίε ορεικτών καυσίμων, αν δεν τι αποκλείσουμε ρητά. Και αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει αξιοπιστία, ώστε το χρήμα να επενδυθεί στην ε, ε, βιωσιμότητα. Δεν θα γίνει όμω εάν υπάρξει το λεγόμενο greenwashing, δηλαδή να τα βάψουν πράσινα ας πούμε και να προσπαθήσουν να τα πουλήσουν ολόκληρο τότε το ε, σχέδιο αυτό για την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση θα καταρρεύσει. Επ' αυτού, αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα σημειώσουμε ως ε, κίνδυνο και θα δούμε αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μέσω της πράσινης ταξονομίας για να εξασφαλίσουμε ότι η πράσινη ταξονομία δεν θα μπει σε τέτοιου είδους ε, τομείς. Σημειώνω το σχόλιο σας και νομίζω ωστόσο ότι ακολουθούμε τους ίδιους στόχους. Κύριε Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, σε λίγες ώρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά του θα εγκρίνει ένα ψήφισμα για τα μεγάλα σκάνδαλα φοροδιαφυγής ΚΟΥΜΕΞ και ΚΟΥΜΚΟΥΜ ζητώντας φορολογική αναρμόνιση, υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών, ισχυροποίηση των ελεγκτικών θεσμών και κυρώσεις για αυτούς που έκλεψαν 55 δισεκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον από τα δημόσια ταμεία επιβαρύνοντας τους συνεπείς φορολογουμένους. Ξέρω ότι η Κομισιόν έχει τις ίδιες προτάσεις. Μας τις ανέπτυξε τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια ο κ. Μοσκοβισή. Πιστεύετε ότι στο Συμβούλιο υπάρχει πολιτική βούληση να κάνουμε αυτά τα βήματα. Το δεύτερο θέμα αφορά την ανάγκη να ολοκληρώσουμε επιτέλους την ε, τραπεζική ενοποίηση με τον τρίτο πυλώνα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και να προχωρήσουν παράλληλα χωρίς καθυστερήσεις και η οδηγία και ο κανονισμός για τα non-performing loans, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχει πολιτική βούληση, στην Κομισιόν υπάρχει, στο Κοινοβούλιο υπάρχει. Στο Συμβούλιο υπάρχει πολιτική βούληση ή θα αναβληθεί και πάλι το θέμα. Και μια τρίτη ερώτηση. Η Κομισιόν παρέχει στήριξη και με δικές σας δηλώσεις στον προϋπολογισμό της χώρας μου, της Ελλάδας για το 2019. Είπατε ότι υπεραποδίδει η ελληνική οικονομία και ε, θα υλοποιήσει τους στόχους της το 2019. Με βάση αυτό θεωρείται εφικτή ναι. σύμφωνα με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα ναι. και την απόφαση του Eurogroup την επιστροφή τη συμφωνημένη της πρώτης δόσης των ελληνικών ομολόγων, κύριε Αντιπρόεδρε, μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2019, όπως έχετε συμφωνήσει και δηλώσει και ο ίδιος. Ε, ε, um, Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν ε, έπιασα όλες τις αποχρώσεις αυτών που είπατε, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω πάντως σε αυτά που θέσατε. Πρώτον, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, ρωτάτε για την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις φορολογικές υπηρεσίες, αν ανταλλάσσουν υπηρεσίες μεταξύ τους. Θα ήθελα λοιπόν να πω επ' αυτού ότι έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και την καταπολέμηση της φοροαπάτης, της διάβρωσης φορολογικής βάσης. Από την πλευρά μάλιστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε να συνεχίσουμε και να δραστηριοποιούμαστε πολύ σε αυτό το τομέα. Πολλά μένουν να γίνουν. Υπάρχουν πολλές σχετικές προτάσεις στο πλαίσιο αυτό, τις οποίες και συζητούμε. Σίγουρα το IT System, το CCTB, την πρότασή μας για το Digitax. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, είναι σαφές ότι στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι μεγάλες ε, εταιρείε, οι πολυεθνικές, πληρώνουν τους φόρους τους. Και δουλεύουμε εντατικά πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια, με ρωτήσατε για το EDIS την εγγύηση καταθέσεων. Εδώ υπάρχει αργή πρόοδος, είναι αλήθεια. Είναι μια νομοθετική πρόταση ήδη του 2015 και δεν προχωρήσαμε πολύ. Από πλευρά του Συμβουλίου τώρα ελπίζουμε να δούμε περισσότερη πρόοδο το Δεκέμβριο στη διάσκεψη κορυφής και την διάσκεψη του Ευρώ γιατί θα τα συζητήσουμε και αυτά τα θέματα για την τραπεζική ενοποίηση, για το MSS, για το EDIS και πιστεύουμε ότι έτσι θα ξέρουμε πόσο πολύ μπορούμε να προχωρήσουμε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπα και εισαγωγικά, πιέζουμε να προχωρήσουμε. Από πλευρά του Κοινοβουλίου περιμένουμε την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής για το EDIS, οπότε η δουλειά πηγαίνει αργά και από τις δύο πλευρές των συνομοθετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως εξακολουθεί να έχει το θέμα στην ημερήσια διάταξη και ελπίζουμε το Δεκέμβριο να έχουμε περισσότερη πρόοδο. Τώρα για τον προπολογισμό 2019 της Ελλάδας. Όσον αφορά τον προπολογισμό αυτό, βλέπουμε ότι τα πράγματα προχωράνε. θα ανταποκριθεί στους στόχους του 3,5% του ΕΠ και σίγουρα θα υπάρξει και φορολογικό περιθώριο και θα μπορέσει η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει ότι χρειάζεται για να μην υπάρξουν οι περικοπές ε, συνταξιδιωτικές. Είμαστε ανοιχτοί σε αυτό. Θα δούμε, πρέπει να υπάρξει διάλογος με τους πιστωτές, ώστε αυτή η προσέγγιση να μπορέσει να λειτουργήσει εφόσον η Ελλάδα αποκρίνεται στους στόχους και στις μεταρρυθμίσεις που αποτελούν και προϋπόθεση για τέτοια μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εσείς ε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπή, Έρχομαι σε έναν τομέα τον οποίο θίξατε προηγουμένως, τα κρυπτονομίσματα και την, ε, τις αρχικές προσφορές ε, νομισμάτων που είναι σημαντικές για την οικονομία και παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο. Και είπατε ότι τον επόμενο μήνα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αναμένουμε ένα regulatory mapping, μια χαρτογράφηση δηλαδή. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι σαφές εάν οι τρέχοντες ορισμοί των χρηματοπιστωτικών εργαλείων, εθνική και ευρωπαϊκή, καλύπτουν τα κρυπτονομίσματα και εάν οι υφιστάμενες διατάξεις, δηλαδή το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, τα καλύπτει επίσης. Μόνο η Παγκόσμια Τράπεζα έχει δώσει συγκεκριμένους ορισμούς και γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω εάν θα λάβετε τους ορισμούς αυτούς ως υποδείγματα για την ε, νομοθετική ρύθμιση στην πρόταση την οποία θα μας καταθέσετε τον ε, Δεκέμβριο. Και ένα δεύτερο, δύο μάλλον, πάλι για τα κρυπτονομίσματα, το ζήτημα της ε, ε, τη της βολατήρης, της αστάθειάς τους δηλαδή. Αν δείτε δηλαδή την κεφαλαιοποίησή τους, έχει ένα μείον 58%, δηλαδή πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. 120 δισεκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Δείχνει πόσο ασταθή είναι ο τομέα αυτό. Και επίση για τη διαφάνεια των κρυπτονομισμάτων, που σήμερα πλέον έχουν ένα ενδιαφέρον για του επενδυτέ λόγω τη ανωνυμία Και μέσα στα πλαίσια της πέμπτη οδηγία για το ξέβλημα βρώμικου χρήματο έχουν ρυθμιστεί, αλλά μερικώ μόνο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν εάν θα λάβετε υπόψη και αυτά τα στοιχεία, δηλαδή αστάθεια και διαφάνεια, αν θα μπουν δηλαδή στη νέα σα νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Έχετε θίξει πλέον πτυχές. Πρώτα για το regulatory mapping. Αυτό κάνουμε τώρα. Ρυθμιστική χαρτογράφηση δηλαδή. Αναμένω έκθεση από τις εποπτικές αρχές και ο στόχος είναι να ανταποκριθούμε σε αυτό ακριβώς το θέμα. Να απαντήσουμε στο ερώτημα δηλαδή, εάν μπορούμε να εφαρμόσουμε την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία ή μήπως χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία κομμένη και γραμμένη ακριβώς για τα κρυπτονομίσματα και τις Αρχικέ προσφορέ. Καθώς επίση για να μπορέσουμε να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στα διάφορα κρυπτονομίσματα και στις αρχικές προσφορές. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά η υποκρυπτόμενη οικονομική δραστηριότητα είναι διαφορετική. Γι' αυτό το λόγο γίνεται η ρυθμιστική χαρτογράφηση. Τώρα για την αστάθεια volatility, που είναι βεβαίως δυστυχώς ένα από τα χαρακτηριστικά των κρυπτονομισμάτων. Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή έχει επικαιροποιήσει τις προειδοποίησεις που εκδίδει για τους επενδυτές ήδη από τον Φεβρουάριο και τονίζει ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου στις επενδύσεις, όπως για παράδειγμα, στις επενδύσεις στα κρυπτονομίσματα εννοείται, όπως η σημαντική αστάθεια, επίσης ότι δεν μπορεί να ορίσει κανείς την προσφορά και ζήτηση και υπάρχει επίσης πάρα πολύ ε, έντονο κερδοσκοπικό στοιχείο και μπορεί κανείς να απολέσει τις επενδύσεις του. Τώρα για το anti-money, ε, anti, μάλλον για τις ε, διατάξεις κατά του ξεπλήματος του χρήματος και αν αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στα κρυπτονομίσματα. Αυτά καλύπτονται από τις απαιτήσει της ε, νομοθετικής ρύθμισης για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Ο κύριος Χόκμαρκ. Ζητώ συγγνώμη, ε, κύριε Ντομπρόφσκης, πρέπει να μεταβώ στην Ολομέλεια λόγω της ε, συζητήσεως για το Brexit εκεί. Θα δώσω όμως την διεύθυνση της συζητήσεως στην ε, κυρία Περβάνου Μπερές. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Μια πολύ σύντομη ερώτηση έχω. Τώρα έχουμε πάνω κάτω ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσει για τα διάφορα τμήματα του τραπεζικού πακέτου και στη διάρκεια αυτών των συζητήσεων Μιλήσαμε για ανώτατα όρια, για ποσοστά, για διαφορές μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν αν σε αυτό το σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα που μας έχουν απασχολήσει αυτά τα νομοθετικά ε, θέματα και πακέτα, εσείς πώς βλέπετε την εικόνα του εισμείωσης του κινδύνου στον τραπεζικό τομέα και στην Τραπεζική Ένωση. Αν αφήσουμε τη συζήτηση για τις διαφορές ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις πίσω μας, τώρα δεν αληθεύει ότι είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από ότι παλιότερα με τη συμφωνία TILAC που περιλαμβάνεται στην BRD καλύτερες και σαφέστερες απαιτήσει για τα κεφάλαια εποπτεία. Θέλετε να μας πείτε πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτή την προοπτική της μείωσης του κινδύνου. Ευχαριστώ, Γκουνάρ, αγαπητοί συνάδελφοι, για τη γενική πρόοδο στην μείωση του κινδύνου. Είναι αλήθεια ότι έχουμε σημειωθεί μεγάλη πρόοδο στη μείωση του κινδύνου τα τελευταία χρόνια και η χθεσινή έκθεση για την Τραπεζική Ένωση που περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το αποδεικνύει αυτό σαφά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν κατέβει κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες δηλαδή 3,4% τώρα. Ε, τώρα, ε, για... Εφάλαμε και τροφυλακτήρες, buffers, ε, που πιστεύω ότι επίσης βοηθούν για τη μείωση του κινδύνου. Έχουμε το backstop για το ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Και όσον αφορά τη συμφωνία για την τραπεζική δέσμη, ε, έχουμε, ε, ε, καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα και τονίζουμε την ανάγκη να ολοκληρωθεί γρήγορα γιατί κάποιες από αυτές τις προδιαγραφές, όπως ας πούμε η πλήρης απώλεια της δυνατότητας εποπτείας, θα πρέπει να ξεκινήσουν να ισχύουν από το επόμενο χρόνο γιατί είναι αυτή η διεθνής μας δέσμευση. Είναι σημαντικό λοιπόν να ολοκληρώσουμε σύντομα όσον αφορά όλες αυτές τις απαιτήσει. Ευχαριστώ. <clears throat> Αυτό σημαίνει δηλαδή ε, μοιρασιά του κινδύνου, κατανομή του κινδύνου. Ο κύριο Βίλκστρομ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Προς το παρόν έχουμε διαπραγματεύσεις που γίνονται για τη ρύθμιση όσον αφορά τις διασυνοριακές ε, πληρωμές. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής και θέλω λοιπόν κύριε Ντομπρόφσκης να σας ρωτήσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει σήμερα στην πράξη για να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια συμφωνία φιλική απέναντι στο χρήστη πριν από τα τέλη της θητείας. Αν επιτρέψετε το χάος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την μετατροπή των νομισμάτων, ε, τότε το αποτέλεσμα είναι οι πληρωμές να γίνονται πιο ακριβές για τον καταναλωτή. Μα ο καταναλωτής, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να ε, υπολογίσει, να συγκρίνει τις τιμές και να ξέρει πού θα πάει. Θέλω λοιπόν κύριε Ντομπρόφσκη να σας ρωτήσω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μόνο δύο προτάσεις ενώ υπάρχουν στο πρόγραμμα δράση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τους ιδιώτες ένα σωρό εναλλακτικέ. Αναφέρεται ότι όλες αυτές οι προτάσεις περιμένουν μέχρι τα τέλη του 2018. Ωραία, θα έχουμε παραπάνω προτάσεις πριν από τα τέλη της θητείας μας. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, χρειάζεται ένα πανευρωπαϊκό σύστημα για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση έτσι ώστε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες να προσφέρονται πιο εύκολα διασυνοριακά με περισσότερο ανταγωνισμό και μείωση των τιμών. Πότε θα υπάρχει μια τέτοια νομοθετική πρόταση από εσά. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές. Ε, φυσικά και χαιρόμαστε για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τους συνομοθέτες στο φάκελο αυτό. Από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε και εμείς να ολοκληρωθεί σε αυτήν τη θητεία αυτός ο φάκελος και διευκολύνουμε όσο μπορούμε το έργο των συνομοθετών από την πλευρά μας. Κάτι το οποίο μας απασχολεί κάπως είναι το εξής. Εμείς προτείνουμε παράταση των τελών των εθνικών σε όλες τις διασυνορικές πληρωμές ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα μιλάει για όλα τα νομίσματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει υποδομή αυτή τη στιγμή που να μπορεί να επιτρέψει να το κάνουμε αυτό με οικονομικά αποδοτικό τρόπο τράπεζες είναι αυτές που περνάνε το βάρος στον καταναλωτή για τις συναλλαγές τώρα, δεν ξέρω, σε σλότι ας πούμε από την Ισπανία στη Βουλγαρία. Δεν υπάρχει υποδομή έτοιμη, η τράπεζα το κάνει και το θέμα είναι αν θα το κάνει με απώλεια ή δεν θα προσφέρει αυτή την υπηρεσία καθόλου. Αυτό είναι που μας προβληματίζει. Και βέβαια θέλω να ε, ξαναπώ ότι το ευρώ θέλουμε να είναι και θα είναι πολύ σύντομα το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, οπότε όταν καταφέρουμε να το πετύχουμε αυτό δεν θα τίθεται ζήτημα. Πάντως θέλω και εγώ να προχωρήσουμε σε αυτό και να το ολοκληρώσουμε γιατί είναι σημαντικό για τους καταναλωτές. Τώρα γιατί μετατροπή των νομισμάτων. Και εδώ κάνουμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις διαφάνειας. Χρειάζεται λίγος χρόνος ώστε τα τερματικά να προσαρμοστούν, να υπάρξει και ένα κάπινγκ, ώστε να μην χρεώνονται υπερβολικά οι καταναλωτές. Συμφωνώ για αυτό που λέτε για τη μετατροπή των νομισμάτων. Έχουμε πρόβλημα εξού και η πρότασή μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε πάνω στις ιδέες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Για τις λιανικές συναλλαγές και το πρόγραμμα δράσης. Αναφερθήκατε στους ελέγχους ψηφιακής ταυτότητας υπάρχουν ομάδες εμπειρογνωμόνων για να δουλέψουν γι' αυτό το ζήτημα και να διασφαλίσουν ότι οι έλεγχοι αυτοί θα χρησιμοποιούνται ευρύτερα. Ένα από τα πράγματα που ήδη κάνουμε είναι ότι έχουμε αφαιρέσει αυτόν τον ε, έλεγχο ως επιπλέον παράγοντα κινδύνου σε σχέση με τη φυσική παρουσία γιατί θεωρείται ότι είναι πιο επικίνδυνες οι ψηφιακές συναλλαγές. Αν αυτό παραμένει ως ιδέα, καταλαβαίνετε ότι δύσκολο θα προωθηθούν οι ψηφιακές συναλλαγές. Πρόεδρος, ωραία, ολοκληρώθηκε εδώ διαρθρωμένος μας ο διάλογος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ που μας παρουσιάζει τον ε, σχεδόν ε, τελικό απολογισμό του έργου σας, μια που πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας μας. Σίγουρα αφήνεται σημαντική κληρονομιά στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επόμενη συνεδρίασή μας είναι κοινή με την Επιτροπή Προϋπολογισμών τη Δευτέρα 3 του μηνός στις 4 μετά μεσημβρίας. Και ο επόμενος η επόμενη ανταλλαγή μαζί σας θα είναι στις 10 Δεκεμβρίου με τον Επίτροπο Μοσκοβισή επίσης. Οπότε θα τα ξαναπούμε τότε. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων που πιστεύω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ.